Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες σήμερα όπου 760 περίπου εκατομμύρια Ευρωπαίοι εκλέγουν πάνω από 700 ευρωβουλευτές. Σας προτείνουμε μια ειδική εκπομπή η Ευρώπη μπροστά στην κρίση. Τι είναι η Ευρώπη, είναι πλεονέκτημα, είναι ελάττωμα, είναι εμπόδιο. Έχουμε λοιπόν εδώ την Καρολίν de Καμαρέ από την France 24, όπως επίσης και τον εκπρόσωπο του Radio France International, του RFI. Έχουμε μεγάλους πρωταγωνιστές της πολιτικής και οικονομικής ζωής. Ο Ιωακή Μαλμούνια, είστε ο Ερπίτροπος, ο αρμόδιος για τα οικονομικά και νομισματικά θέματα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ζωηρή, έτσι δεν είναι. Μόνο για οικονομία μιλάμε, είναι αλήθεια λέει ο Αλμούνια. Κυρία Φαϊμπέργα, σας καλωσορίζω. Ήσασταν πρόεδρος της Λετωνίας, είστε αντιπρόεδρος της ομάδας των σοφών, οι οποίοι ασχολούνται με το ρόλο της Ευρώπης στον ορίζοντα του 2030. Είστε η καλύτερη πρέσβυρα της δικής σας χώρας. Σίγουρα καλώς ήρθατε από τη Ρήγα. Έχουμε επίση μαζί μα και την Νικόλ Φοντέν. Ήσασταν υπουργό στην γαλλική κυβέρνηση, ήσασταν και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1999 μέχρι το 2002. Εγκαταλείπετε το κοινοβούλιο αφού περάσατε εδώ πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε και δύο δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. Έχουμε τον David Ρένι από τον Economist και την Zetnik από την Σλοβενική τηλεόραση. Να πω στους ε, τηλεθεατές ε, ε, της France 24 όπως επίσης και στους ακροατές ε, του RFE ότι έχουμε προβλήματα γιατί ε, υπάρχει μια προσπάθεια έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των εκπομπών του RFE International, του Διεθνούς Γαλλόφωνου Ραδιοφώνου, ιδιαίτερα όταν εκπέμπει σε άλλες γλώσσες όπως τα αλβανικά, τα σουηδικά κτλ. Πάση περιπτώσει, α μιλήσουμε για τη συμμετοχή στι εκλογέ. Κυρία Φοντέν, από ό,τι φαίνεται η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Γιατί δεν ενδιαφέρονται οι πολίτε για την Ευρώπη, κυρία Φοντέν. Είναι αλήθεια ότι οι πολίτε δεν συνειδητοποιούν πραγματικά τον σημαντικό ρόλο που παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι αλήθεια ότι η αύξηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν σταδιακή. Από τη μία ξεκινήσαμε με την καθολική ψηφοφορία, μετά με την συναπόφαση μέσω της συνθήκης του Μάστριχτ γιατί συναποφασίζουμε με το Συμβούλιο Υπουργών. Και συγγνώμη κύριε Υπουργέ, θα έλεγα ότι από το ε, 1999 ανατρέψαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό ήταν μια ιδρυτική πράξη θα έλεγα σημαντική πολιτικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Ιωακή Μαλμούνια, είστε ο Ευρωπαίο Επίτροπο, ο υπεύθυνο για τα οικονομικά θέματα. Ασχολείστε με την οικονομική κρίση. Ανησυχεί ο πολίτη για την ανεργία, για τη μείωση της καταναλωτικής σου δύναμης. Είδαμε κάποια προγράμματα ανάκαμψης, αλλά τελικά η αντίληψη που κυριαρχεί είναι ότι η Ευρώπη δεν είναι εδώ, είναι απούσα η Ευρώπη, κάνει κάτι η Ευρώπη. Κοιτάξτε, Ίσως να υπάρχει ένα θέμα πληροφόρησης γύρω από τα ευρωπαϊκά θέματα, λέει ο κύριο Σαλμούνια. Ήδη από τον Νοέμβριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ένα πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης το οποίο ενέκριναν και το οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζουν, το οποίο υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη παράγει αποτελέσματα θετικά. Συνέπεια αυτή τη ευρωπαϊκή δράση είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάρχει υπάρχει μια τόσο σημαντική οικονομική απόφαση από κοινού, βλέπουμε ότι οι επιπτώσεις μέσω της δημοσιονομικής στήριξης της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι στο ίδιο ύψος περίπου με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δική σας χώρα, η Ισπανία η Αλμούνια, όπως επίσης και η δική σας χώρα, η Λετωνία, αναγκάστηκε να δανειστεί 7 δις ευρώ Κυρία Φραϊμπέργα, κάποια χρόνια μετά την ένταξη, μήπως η Λετωνία θεωρεί ότι δεν βοηθήθηκε ιδιαίτερα από την Ευρώπη. Νομίζω ότι η κρίση χτύπησε τη Λετωνία με πάρα πολύ απότομο τρόπο. Κανένας φυσικά δεν μας προειδοποίησε, αυτό είναι αυτονόητο. Ταυτόχρονα η χώρα θα ήθελα να πω ότι ακολουθούσαμε θα έλεγα ένα αριθμό ανάπτυξης ηλικιώδη και αυτό δεν ήταν απόλυτα θετικό. Γι' αυτό και μας χτύπησε η κρίση. Οι διαδικασίες άλλαξαν πάρα πολύ γρήγορα και δυστυχώς συνεχίζουν να είναι αρνητικές. Γι' αυτό ακριβώς αυτό το πρόγραμμα ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κεφαλαιόδη μα σημασία. Νομίζω ότι για τον πληθυσμό μας, για τους πολίτες μας θα δώσει εμπιστοσύνη στους πολίτες, θα δώσει εμπιστοσύνη αυτό το πρόγραμμα στους επενδυτές και θα σταθεροποιηθεί σε κάποια στιγμή η κατάσταση. Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κρίσιμη και δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντική. Κυρία Φοντέν, συμφωνείτε, υπάρχει η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη απέναντι στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Μήπως κάποιοι τη θεωρούν ανεπαρκή Κοιτάξτε, η αλληλεγγύη αυτή σίγουρα δεν είναι επαρκή. Είναι σαφέ ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Αλλά να πω στον κύριο Επίτροπο κάτι το οποίο γνωρίζει καλά βέβαια. Δεν κατανοήσαμε ότι έρχεται η οικονομική κρίση. Αλλά πριν την κρίση η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έθετε το θέμα του ελέγχου των χρηματαγορών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ξέρετε κύριε Αλμούνια. Έχουμε ανταλλάξει απόψεις πάρα πολλές φορές. Και θα έλεγα ότι εμείς δημιουργήσαμε την ομάδα του Ζακ de Η ομάδα αυτή κάνει μια εξαιρετικά χρήσιμη δουλειά. Ελπίζω τα αποτελέσματά της να χρησιμοποιηθούν με σωστό τρόπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αλληλεγγύη ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη κυρίες και κύριοι. Είναι σαφές ότι αποφύγαμε μια μεγάλη πιστοτική ευρωπαϊκή κρίση, τραπεζική κρίση, η οποία θα είχε δραματικά, μα δραματικά αποτελέσματα. Και στα πλαίσια της ομάδας το 20, της ομάδας των 20 λοιπόν, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να ελεγχθεί ο διεθνής χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός. Να μου επιτρέψετε να θυμίσω επίσης τον ρόλο τον οποίο έπαιξε το ευρώ. Δεν το υπογραμμίζουμε όσο χρειάζεται αυτό, όσο πρέπει να το κάνουμε. Πράγματι το ευρώ μας βοήθησε έτσι ώστε να αποφύγουμε δραματικές συνέπειες. Αν δεν είχαμε στη διάθεσή μας το ευρώ θα ήμασταν σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη από αυτήν που βρισκόμαστε σήμερα. Συμφωνεί και η κυρία Φραϊμπέργκα. Καλώς. Βλέπω εδώ τον κύριο Ζίτνικ, ο οποίος ε, είναι δημοσιογράφος της Σλοβενικής τηλεόρασης, κρατική τηλεόραση της Λιουμπλιάνα. Έντβαρντ Ζλίτνικ. Έχετε μια ερώτηση προς τον κύριο Αλμούνια να θέσετε. Κύριε Επίτροπε, είμαι βέβαιος ότι η εισαγωγή του ευρώ στη Σλοβενία ήταν επιτυχής και πράγματι βοήθησε να ξεπεράσουμε τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης. Πιστεύετε ότι τα κριτήρια για την ένταξη στη ζώνη ευρώ θα πρέπει να ερμηνευθούν με πιο ευέλικτο τρόπο έτσι ώστε να βοηθηθούν γρηγορότερα κάποιες άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Χώρες θυμίζουν που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Και κυρία Φαϊμπέργα, ίσως και εσείς θα ήθελατε να σχολιάσετε τη δυνατότητα εισόδου ε, στη ζώνη ευρώ. Ο Επίτροπο Αλμούνια, πράγματι είναι μεγάλη επιτυχία το ευρώ και προστατεύει την ευρωπαϊκή οικονομία. 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκουν στην Ευρωζώνη. Αλλά υπάρχουν χώρε που θέλουν να μπουν στη ζώνη αυτή, η Λιθουανία, η Λετωνία και άλλε. Στην περίπτωση τη Λετωνία, να πω ότι βρισκόμαστε στο στάδιο διαπραγμάτευση του τελευταίου μήνε, σε καθημερινή βάση, με τι λετωνικέ αρχέ. Προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να ξεφύγουμε από αυτή τη δύσκολη κρίση που εν πολλής οι αρχές της χώρας αυτής είχαν προβλέψει. Αυτό το αναγνωρίζω. Δυστυχώς συνέβη αυτό το οποίο συνέβη. Πράγματι το ευρώ βοηθάει τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακριβώς η προσπάθεια της Λετωνίας να ανήκει στην Ευρωζώνη τα επόμενα χρόνια μέσω πρόθεσμα είναι κάτι το οποίο λειτουργεί θετικά και καθιστά ιδιαίτερα συνεκτικές τις προσπάθειες μεταρρύθμισης της λετωνικής οικονομίας. Στην περίπτωση της Λετωνίας, της Ρουμανίας, της Ουγγαρίας νομίζω ότι έχουμε ξεκάθαρο το παράδειγμα της αλληλεγγύης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Η κυρία Νικόλ Φοντέν. Ε, πρέπει να δώσω κάποιου αριθμού, κυρία Φοντέν. Η αλληλεγγύη σαν ιδέα είναι καλή, αλλά ακούγεται κάπω αφηρημένη. Είχαμε ένα ειδικό μέσο για τη χρηματοδότηση, τη εξωτερική χρηματοδότηση των χωρών που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Εδώ και 7 μήνε είχαμε στη διάθεσή μα 12 δι. Σήμερα του θέτουμε στη διάθεσή του 50 δι. Και εμεί το προτείνουμε αυτό. Τετραπλασιάσαμε δηλαδή τους σπόρους τους οποίους μπορούμε να προσανατολίσουμε προς τις ανάγκες των χωρών αυτών. Συνεπώς αυτό αποδεικνύει έμπρακτα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αυτό ακολουθήθηκε από μια αύξηση της ε, οικονομικής δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με μια προκαταβολή των πληρωμών των διαφθορτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής μια στενή συνεργασία με τη Λετωνία και την Ουγγαρία για να βοηθήσουμε τι μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται οι χώρε αυτέ. Κυρία Φραϊμπέργα, ακούσατε αυτά τα οποία ισχυρίζει το Επίτροπο Σαλμούνια, είστε ικανοποιημένοι τελικά. Μήπω περιμένετε περισσότερα από την Ευρώπη. Μια οικονομική διακυβέρνηση. Θέλετε να ενταχθεί πραγματικά η χώρα σα στην Ευρωζώνη. Ένα ευρωδάνειο και τα ευρωμόλογα σα φαίνονται ελκυστικά. Εγώ λυπάμαι που η χώρα μου δεν μπόρεσε να σεβαστεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα που θα τη είχε επιτρέψει να είναι ε, την 1η Ιανουαρίου του 2008 στη ζώνη ευρώ. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίσαμε πραγματικά να αυξάνουμε με κάποιο τρόπο ανεξέλεγκτο θα έλεγα τον πληθωρισμό. Και αυτός ο ρυθμός δεν μας επέτρεψε να σεβαστούμε τα κριτήρια για την ένταξη στη ζώνη ευρώ. Αυτό ήταν δυστυχές για τη χώρα μου. Γιατί οι υπόλοιποι μακροοικονομικοί δείκτες, εκείνη την εποχή τουλάχιστον, ήταν πραγματικά αυτοί που χρειάζονταν. Αλλά δυστυχώς το θέμα του δείκτη του πληθωρισμού δεν μας επέτρεψε και η κυβέρνηση δεν ήταν εν πάση περιπτώσει σε θέση να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό. Δεν είχε τα μέσα που χρειαζόταν στη διάθεσή της. Από τη μία υπήρχαν τα διαφορετικά ταμεία, τα οποία χρηματοδοτούσαν τις αγορές. Υπήρχαν πάρα πολλοί πολίτες της Λετωνίας που εργαζόντουσαν στο εξωτερικό και έστελναν συνάλλαγμα, ευρώ δηλαδή στη χώρα μου. Υπήρχε μια εσωτερική κατανάλωση η οποία αυξανόταν αλόγιστα. Αυτό οδήγησε σε αύξηση των τιμών λιανικής Υπήρξε και μια αύξηση των πόρων προερχομένων από την παραγωγή ενέργειας. Όλα αυτά έπαιξαν ρόλο συνδυαστικά. Και τώρα πια τα δύσκολα έχουν έρθει και είναι πολύ πιο δύσκολα θα έλεγα από ό,τι στο παρελθόν. Η κυρία Νικόλ Φοντέν, θα ήθελα να υπενθυμίσω εδώ κάτι. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κάποια δημοσιονομικά μέσα τα οποία χαρακτηρίζω ανεπαρκή, ανεπαρκέστατα και δεν είναι στο ύψος των φιλοδοξιών μας σε επίπεδο πολιτικό. Πράγματι θα πρέπει να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό δάνειο. Κοιτάξτε, θα πρέπει να επανεξεταστεί η μέθοδος λειτουργίας η δημοσιονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι το συζητάμε εδώ και χρόνια το θέμα αυτό. Βλέπετε οι Ηνωμένε Πολιτείε μετά από την κρίση του 1929 άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. 70 χρόνια εμείς μετά, εμείς στην Ευρώπη δεν πήραμε τα κατάλληλα μαθήματα. Εγώ θα ήθελα να αλλάξουν τα πράγματα. Θέλω ένα ευρωπαϊκό New Deal. Πράγματι η Ευρώπη, λέει ο Χωακή Μαλμούνια, έχει ανάγκη από ένα ισχυρότερο προπολογισμό. Δυστυχώ όμω οι κυβερνήσει των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι οι αρμόδιε επί του προπολογισμού αρχέ, δεν το έχουν επιτρέψει. Δεν έχουν ακολουθήσει τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι οποίε έκανε εδώ και πέντε χρόνια. Πάντω, για να βοηθήσουμε μια χώρα συνεχίζει ο Επίτροπος σαν τη Λετωνία σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία, όπως είπα, τετραπλασιάσαμε την οικονομική βοήθεια. Τετραπλασιάσαμε σε λίγους μήνες. Αυτό δείχνει ότι είμαστε σε θέση να δανειστούμε χρήματα όταν δεν τα έχουμε για να βοηθήσουμε τη Λετωνία. Εγώ είμαι υπεύθυνο, γι' αυτό βγαίνω στην αγορά και βρίσκω χρήματα για να βοηθήσω. Τα τελευταία πέντε δις που δώσαμε στις χώρες αυτές, Ουγγαρία, Ρουμανία, Λετωνία, προσφύγαμε στις χρηματαγορές σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, εγώ δεν μιλάω για πέντε δις, ένα μεγάλο, εν πάση περιπτώσει, ευρωδάνειο, χιλίων δις ίσως, για τις τεχνολογίες, για την έρευνα και την ανάπτυξη. Ναι, ναι. ναι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τέτοια είδου μέσα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, λέει ο επίτροπο αύξησε κατά 30% την δανειοδοτική της ικανότητα. Τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στέλνουν ποσά, πόρους προς χώρες όπως η Λετωνία και η Ουγγαρία 4% περισσότερα κάθε χρόνο. Πρέπει να ενισχύσουμε επίσης και τη δυνατότητα απορρόφησης των ποσών αυτών από τις συγκεκριμένες χώρες. Θα πρέπει να βοηθάμε τις χώρες αυτές να απορροφούν τα χρήματα και να δαπανώνται τη συγκεκριμένη πόρη. Αν πείσουμε τον Ευρωπαίο πολίτη ότι θα πρέπει να προσπαθήσει να κατανοήσει το πόσο χρήσιμη είναι η Ευρώπη, να ψηφίζει για την Ευρώπη. Αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να του εξηγήσουμε τι κάνουμε. Κάνουμε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε εδώ και πέντε χρόνια ήταν επιτυχής. Κύριε Επίτροπε έχετε δίκιο λέει η κυρία Φοντέν. Αύριο όμως εσείς θα υποστηρίξετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν αυτό αποφασίσει να ζητήσει την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Να υπάρξουν νέα δημοσιονομικά μέσα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως λέει ο Επίτροπος Σαμούλια. Πράγματι εγώ σαν Επίτροπος εδώ και πέντε χρόνια όταν συζητούσαμε μαζί σας τις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007 με 2013 είδα ότι και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησαν ποσά που ήταν πολύ λιγότερο φιλόδοξα από αυτά τα οποία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά εγώ πιστεύω στην Ευρώπη. Όλοι πρέπει να πιστεύουμε στην Ευρώπη. Όσοι είμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το κάνουμε αυτό. Το θέμα είναι ποια είναι τα βήματα τα συγκεκριμένα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε σε καθημερινή βάση για να στηρίξουμε την Ευρώπη. Πράγματι για να στηρίξουμε την Ευρώπη λέει η κυρία Φοντέν πρέπει να έχουμε τα μέσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυρία Φαϊμπέργα, ο κύριος Επίτροπος είπε ότι οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα μου θα πρέπει να συνεχιστούν. Βεβαίως και θα πρέπει να συνεχιστούν. Είμαι σίγουρος ότι ακόμα και σήμερα αυτή την ώρα δουλεύουν γι' αυτό. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω ότι στο πρόγραμμα βοήθειας προς τις νέες χώρες μέλη πρέπει κάτι να υπογραμμίσω. Θα πρέπει να επωφεληθούμε από την παρούσα κρίση, έτσι ώστε να βρούμε τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους διανέμονται τα ποσά αυτά και βρίσκουν τους σωστούς παραλήπτες. Στην Λετωνία θα έλεγα υπάρχει κάτι το οποίο δυσκολεύει την κατάσταση. Υπάρχει μια τροχοπέδη στην ταχύτητα με την οποία μπορούν τα χρήματα αυτά να προχωρήσουν. Mm. Υπάρχει πράγματι μια δυσκινησία, μια γραφειοκρατική επιβάρυνση. Σε επίπεδο μεθοδολογικό λοιπόν, σε επίπεδο διαδικασιών πρέπει να απλουστεύσουμε πάρα πολλά πράγματα. Οι πολίτες, οι Λετονοί παραπονούνται γι' αυτό. Βλέπουν ότι έχουν ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα. Δανείζονται χρήματα για να αυτοχρηματοδοτήσουν κάποιες αγορές για να προχωρήσει το πρόγραμμά mm. τους mm. περιμένουν πάρα πολύ καιρό για να πάρουν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στην απορρόφηση των συγκεκριμένων ποσών. Να επιτρέψτε μου να πω κάτι εδώ λέει ο κύριος Σαλμούνια οι χώρες δεν έχουν την ίδια απορροφητική ικανότητα. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες πρέπει να κάνουν περισσότερα. Και αυτό εξαρτάται από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές της κάθε χώρας. Πράγματι δεν χρειάζεται η γραφειοκρατία να καταστρέφει αυτά τα προγράμματα. Έχετε δίκιο. Και ένας λόγος είναι ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των προγραμμάτων αυτών είναι σκληρός εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια κάθε χώρα έχει διαφορετικούς ρυθμούς απορρόφησης. Κάποιες χώρες τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα από άλλες. Πρέπει να δούμε λοιπόν το είδος της μεταρρύθμισης το οποίο απαιτείται. Να δούμε πώς θα προσανατολίσουμε τις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις. Μια χώρα σαν τη δική σας πρέπει να συγκλίνει προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συνεπώς οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι μόνο τέτοιου είδους που απαιτούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Κάποιες χρηματοδοτήσεις πρέπει να αποφασίζονται και να εκτελούνται θα έλεγα με την πολιτική συνένεση και την κοινωνική συνένεση στην συγκεκριμένη χώρα και μόνο. Υπάρχουν παραδείγματα επιτυχίας. Υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες δεν τα κατάφεραν τόσο καλά. Με τους ίδιους κανόνες, με τις ίδιες διαδικασίες τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Λοιπόν, θα πρέπει να βοηθήσει η Ευρώπη. Η Ευρώπη κατανοεί αυτή τη στιγμή τα προβλήματα, τις φιλοδοξίες, τις δυσκολίες των νέων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πούμε και εμείς σαν Ευρώπη στους υπευθύνους τους πολιτικούς των χωρών αυτών ότι πρέπει να κάνουν και αυτοί την δική τους προσπάθεια. Πράγματι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το μέγεθος των προγραμμάτων αυτών. Ο εκπρόσωπος του Economist. Σας ακούω, παρακολουθείτε και βράζετε λιγάκι και θα θέσετε ένα ερώτημα το οποίο είναι διαφορετικό από αυτά τα οποία ακούμε. Εσείς έχετε μια σελίδα στο Economist η οποία ονομάζεται Καρλομάγνος, Ε, Είστε πάντα υπέρ της φιλελεύθερης αντίληψης για την αγορά. Κοιτάξτε, να θέσω ένα ερώτημα. Ακούμε πάρα πολλά πράγματα για την Ευρώπη, για περισσότερη Ευρώπη κτλ. Λες και η Ευρώπη είναι ένας μηχανισμός που παράγει χρήμα και θα βελτιώσει τη λειτουργία των οικονομιών μας. Εγώ πίσω από αυτά βλέπω μια συγκεκριμένη ιδεολογική αντίληψη για την Ευρώπη. Μια Ευρώπη υπερδιακανονιστική του χρηματοπιστωτικού τομέα. Όταν βλέπω ότι θα πρέπει να απαιτηθούν περισσότερες δυνατότητες για ελέγχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακούω από την Γερμανία να δοθεί προτεραιότητα μικρότερη από ό,τι δίδεται σήμερα στις πολιτικές του ανταγωνισμού στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής. Και αυτό με εκπλήσει εδώ στις Βρυξέλλες. Κατηδίαν μου είπαν διάφοροι ανώτατοι υπάλληλοι εδώ στο Κοινοβούλιο ότι κάποιες πολιτικές για μικρότερο ανταγωνισμό, για περισσότερο διακανονισμό, για περισσότερες ρυθμίσεις, για μεγαλύτερους φόρους είναι κάποιες ε, απόψεις οι οποίες κυκλοφορούν πολύ και δυστυχώς δεν θα βοηθήσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης. Βέβαια αυτά τα ακούω στους διαδρόμους και αναρωτιέμαι αν οι πολιτικοί υπεύθυνοι που προωθούν τις θέσεις αυτές είναι σε θέση να είναι ειλικρινείς και να πούνε ότι πράγματι θα πρέπει να αλλάξουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αλλά τα πρότυπα αυτά θα οδηγήσουν σε μικρότερους ρυθμούς ανάπτυξης και οι μικρότεροι ρυθμοί ανάπτυξης θα δημιουργήσουν σε λιγότερες θέσεις απασχόλησης. Λοιπόν για να βγούμε από την κρίση τι θέλουμε, θέλουμε περισσότερη Ευρώπη ή λιγότερη Ευρώπη. Πράγματι, ε, το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη παρεμβατικότητα ή όχι στις αγορές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα χρηματοπιστωτικά ας πούμε, πρέπει να υπάρξουν περισσότερες παρεμβάσεις και γι' αυτό καταστράφηκε το σύστημα. Υπήρξαν καταχρήσεις. Πράγματι αυτοί που, ε, ε, οι ίδιοι που εργάζονται στον ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα λένε ότι θα πρέπει να, απαιτηθ, να απαιτούνται νέοι κανόνες εν πάση περιπτώσει. Πρέπει λοιπόν σε πολλούς τομείς να υπάρξουν παρεμβάσεις. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε προς τον Ευρωπαίο πολίτη, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι οι κανόνες αυτοί, οι νόμοι αυτοί δεν θα πρέπει να πνίξουν τον δυναμισμό της οικονομίας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε την δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερο δυναμισμό, να αυξήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης, μια πραγματική ισχυρή ανάπτυξη βασισμένη, εδρεωμένη στην παραγωγικότητα, στην καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση. Θα πρέπει να τα συνδυάσουμε λοιπόν την οικονομική ανάπτυξη από τη μία και την κοινωνική Ευρώπη από την άλλη, γιατί έχουμε και κοινωνικές αντιλήψεις για την Ευρώπη. Συμφωνώ απόλυτα με την απάντηση του Επιτρόπου Αλμούνια, λέει η κυρία Φοντέν. Αυτό το οποίο έχουμε προτείνει κύριε Επίτροπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον έλεγχο των χρηματαγορών σαν παράδειγμα, για τις ασφάλειες, για τις ε, εταιρείες βαθμολόγησης και αξιολόγησης των εθνικών οικονομιών, είναι πράγματα τα οποία δεν είναι εναντίον των αρχών του ανταγωνισμού. Πρέπει να βρούμε βέβαια κάποιες ευαίσθητες γραμμές ισορροπίας, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ταυτόχρονα ότι το χειρότερο σε αυτή τη φάση θα ήταν κάποιες προστατευτικές πολιτικές. Όχι στον προστατευτισμό. Όλοι συμφωνούμε ότι θα ήταν αρνητικός, δραματικός μάλιστα. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μια διεθνή συνεργασία για να αποφύγουμε αυτές τις προστατευτικές τάσεις. Σαν παράδειγμα, περιμένετε προτάσεις από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα hedge funds. Ακούσαμε την πιθανή πρόταση Μακρύβη, η οποία διευκολύνει την εγκατάσταση των hedge funds στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, εμείς δεν θέλουμε να διευκολύνουμε. Εμείς θέλουμε ίσα ίσα να ρυθμίσουμε να καταγράψουμε και να ελέγξουμε τις δραστηριότητες των hedge funds στην Ευρώπη. Για πρώτη φορά το κάνουμε αυτό. Αυτό ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κοινοβούλιο είναι κάτι ε, το οποίο υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίχθηκε και από την ομάδα των 20 και στι Ηνωμένε Πολιτείε γίνεται ακριβώ το ίδιο σα θυμίζω. Θα πρέπει να μην υπάρχουν οικονομικέ δραστηριότητε και οικονομικά προϊόντα τα οποία να διαφεύγουν κάθε μορφή ελέγχου. Επί τη αρχή, λέει η κυρία Φοντέν συμφωνούμε. Αλλά έχουμε ορισμένε επιφυλάξει και υπάρχουν δύο συγκεκριμένοι κίνδυνοι. Ο πρώτο κίνδυνο είναι να επιτρέψουμε την κυκλοφορία κάποιων οικονομικών προϊόντων από οικονομικού παραδείσου των οποίων οι διαχειριστές θα είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μια δεύτερη παρατήρηση, ένας δεύτερος κίνδυνος βέβαια, είναι ότι αυτό το οποίο πραγματικά επιθυμούμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει κάτι τέτοιο, κυρία Φοντέν, λέει ο Ιωακή Μαλμούνια. Κοιτάξτε, θα πρέπει να τα ελέγξουμε όλα αυτά. Θα πρέπει τα ταμεία αυτά να είναι διαφανή και να είναι εύρυθμη και χρηστή λειτουργία τους. Εγώ δεν θα είμαι πλέον ευρωβουλευτής λέει η κυρία Φοντέν, αλλά αυτή είναι η σωστή πορεία. Κοιτάξτε, εφόσον υπάρχουν τέτοιου είδου ταμεία τα οποία λειτουργούν στην Ευρώπη, προφανώ και θα τα ελέγχουμε. Ποια είναι η κατάσταση όμω. Το θέμα είναι ότι η πλειοψηφία των hedge funds δεν είναι εγκατεστημένα στην Ευρώπη. Ούτε στην υπηρετική Ευρώπη, ούτε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι οι τα νήσου καημάνου καταγεγραμμένα όλα αυτά τα ταμεία. Οπότε τι γίνεται, εμεί τι μπορούμε να κάνουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση για να ελέγξουμε δραστηριότητε σε τέτοιου είδου χώρε. Η κυρία Φαϊμπέργα, κοιτάξτε, ε, υπάρχουν τέτοια ταμεία και στην Ευρώπη. Ας μην κρύβουμε την αλήθεια. Υπάρχουν τέτοια ταμεία ιδιαίτερα ισχυρά σε επίπεδο κεφαλαίου. Λοιπόν, ας ελέγξουμε αυτά τα ταμεία, ας διασφαλίσουμε τη διαφάνεια σε αυτά τα ταμεία. Και αυτό θα είναι ένα καλό παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο. Και θα ε, ενθαρρύνουμε και άλλες κυβερνήσεις εθνικές ή όπως την κυβέρνηση της πολιτείας του Ντέλαγουερ σαν παράδειγμα που είναι τέτοια ταμεία πάρα πολλά καταγεγραμμένα εκεί να βοηθήσουν την εύρυθμη λειτουργία τους. Το θέμα δεν είναι μόνο να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία των ταμείων αυτών για τις επενδύσεις των συνταξιοδοτικών ταμείων. Το θέμα είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Να υπάρξει μια οικονομική ανάπτυξη η οποία να μην είναι τόσο δύσκολη όσο η σημερινή. Αυτή τη στιγμή ψυχολογικά υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες στο επίπεδο κατανάλωσης Υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχουμε αναφερθεί. Ανεργία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό μέσο όρο 10%. Σε κάποιες χώρες έχουμε φτάσει περίπου στο 20% όπως τη Λετωνία. Η κατάσταση ε, πράγματι είναι πολύ επικίνδυνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει ε, επίδειξη θάρρους και φαντασίας και να βρει κάποιες λύσεις. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε λέει ο Ακή Μαλμούνια. Ξεκινήσαμε ορισμένες πρωτοβουλίες με την τσεχική προεδρία. Κάναμε μια συνάντηση κορυφής για την απασχόληση χωρίς πολύ μεγάλη επιτυχία λέει ο δημοσιογράφος. Όχι, γιατί το λέτε αυτό. Ακούστε λίγο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε αυτή τη συνάντηση κορυφής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έλεγα πρότεινε να γίνει αυτή η συνάντηση κορυφής. Οι εθνικοί εταίροι πράγματι ήθελαν να είναι παρόντε και να τα συζητήσουν τα θέματα. Ορισμένες κυβερνήσεις κρατών μελών αφού δακτυλοδεικτούν τις Βρυξέλλες και λένε αυτές φταίνε, όταν οι Βρυξέλλες κάνουν προτάσεις για την ανεργία δεν δέχονται να ληφθούν τέτοιου είδους μέτρα. Είπαμε λοιπόν, ας πάμε όλοι στη συνάντηση κορυφής στην Πράγα και κάποιες κυβερνήσεις εκεί δεν ανταποκρίθηκαν, είπαν ότι έχουμε δουλειά, δεν μπορούμε να πάμε. Ας μην κατηγορούν τις Βρυξέλλες λοιπόν. Καλώς, έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Σε λίγες ώρες θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Κυρία Φαϊμπέργα, τι φοβάστε περισσότερο. Ελπίζω ότι οι προβλέψεις που έλεγαν ότι θα υπερψηφιστούν τα ακραία πολιτικά κόμματα θα διαψευστούν και ελπίζω ότι οι εκλογείς θα κρατήσουν τη λογική που απαιτείται, θα ψηφίσουν ισορροπημένα και δεν θα δώσουμε κέρδη σε ακραία πολιτικά κόμματα. Νικόλ Φοντέν. Φοβάστε ή ελπίζετε. Εγώ θέλω ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανοιχτό στον υπόλοιπο κόσμο ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θέλει να ελέγξει την κρίση αλλά όχι εις βάρος των χωρών του τρίτου κόσμου. Και θυμίζω εγώ ότι έχουμε πολλά θέματα εδώ. Το θέμα της μεταρρύθμισης για μια ακόμη φορά της κοινή αγροτικής πολιτικής, της αηφόρου αναπτύξεως, οικολογικής οικονομικής ανάπτυξης. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν δείχνοντας αλληλεγγύη στον τρίτο κόσμο κλείνει ο κύριος Σαλμούνια. Ελπίζω το νέο κοινοβούλιο που εκλέγεται σήμερα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών. Ένα κοινοβούλιο που να είναι σε θέση να πει στον Ευρωπαίο πολίτη σε καθημερινή βάση το τι συζητάμε, το τι αποφασίζουμε, το τι πετυχαίνουμε. Κλείνει η συζήτηση αυτή. Θα συνεχίσει, θυμίζω, η εκλογική βραδιά. Μείνετε στο κανάλι μας. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας επέτρεψε να κάνουμε αυτή την χρήσιμη κατά τα άλλα συζήτηση.